Γκάλ Erasmus και άλλα εργαλεία για την πρόθεση της κινητικότητας στο πλαίσιο τη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Ο εισηγητή, τέσσερα λεπτά. Η έκθεση αυτή απορρέει από μία έκθεση της Υποεπιτροπής Πολιτισμού και Εκπαίδευσης και συμπληρώνει την εργασία της Επιτροπής Απασχόλησης. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει συμπληρωματικός χαρακτήρας των δύο και θέλουμε να βρούμε στοιχεία θετικής επίλυσης μίας εξίσωσης μεταξύ εκπαίδευσης κατάρτισης και από την άλλη εργασίας για τόσους νέους. Άρα Επίτροπε, βρισκόμαστε πολύ μακριά από τη σωστή οδό για να ανταποκριθούμε στους στόχους που είχαμε εμείς ορίσει μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής 2020. Ε, Φαίνεται ότι αποκλίνουμε κιόλας. Γι' αυτό ακριβώς ε, ζητήσαμε να βελτιωθεί το Erasmus Plus για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην επαγγελματική κατάρτιση. Ορίζουμε λοιπόν τα προσκόμματα που υπάρχουν και τις ανεπάρκειες του Erasmus Plus και ορίζει τους ε, βασικούς άξονες προσαρμογής για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στους ε, επαγγελματικούς στόχους, στους στόχους επαγγελματικής κατάρτισης. Κινητικότητα σημαίνει απασχολησιμότητα και αυτό θα πρέπει να γίνει το γενικό μας γνωμικό. Ελπίζω να μπορέσουμε να αποτανθούμε στην ε, Επιτροπή και στα κράτη-μέλη απαιτώντας ε, συγκεκριμένα μέτρα σύγκλησης. Το θέμα επίγει. Θα πρέπει να ε, βοηθήσουμε και να βελτιώσουμε τις εναλλακτικές λύσεις κινητικότητας και απασχολησιμότητας. Να ισχύσουν συμπληρωματικά μέτρα με προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Επίσης, να χρησιμοποιήσουμε τους κατάλληλους πόρους για να δούμε ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες της επαγγελματικής κατάρτισης. Να άρουμε προσκόμματα για να μπορέσει να επιτύχει αυτό το πλαίσιο. Ε, να ξεπεράσουμε δηλαδή το φράγμα της γλώσσας, των διαφορετικών γλωσσών. Επίσης θα πρέπει να δούμε ποιοι θα είναι οι ενδιάμεσοι φορείς που θα προβάλλουν νέα πρότυπα διαχείρισης του Εράσμου ΣΥΝ. Γι' αυτό να δούμε πώς θα μπορέσουμε να ορίσουμε ε, οργανισμούς ή κοινοπραξίες που θα πρέπει να συμφωνήσουν για να δώσουν τις κατάλληλες απαντήσεις. Θα πρέπει να υπάρξει αλληλοαναγνώριση τίτλων σπουδών, κάτι το οποίο δεν ισχύει πάντα. Θα πρέπει να γίνει πλέον. Και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την έννοια του μαθητευόμενου Ευρωπαίου, όπως ορίζεται στην έκθεση. Αυτό αφορά και τους διδάσκοντες που κατέχουν θέση κλειδί. Θα πρέπει να βρει το Εράσμους ΣΥΝ την πραγματική του θέση σε, αυτή την, σε αυτό το πλαίσιο. Πρέπει να ολοκληρώσετε. Θα πρέπει λοιπόν να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα Εράσμους ΣΥΝ σε αυτά τα πλαίσια. Ευχαριστώ και τώρα πάμε στη διαδικασία Καρστιάη. Έχω πολλοί αριθμές, πολλοί αριθμοί αιτήματα. Θα δώσω σε δύο από το ΕΛΚ και τους σοσιαλιστές και σε έναν ομιλητή από τις λοιπές ομάδες. Ελπίζω να δείξετε και εσείς κατανόηση. Μπότσκορ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για, συγγνώμη τον εισηγητή για ε, ένα έγγραφο πολύ καλή ποιότητα. Η γενετικότητα λοιπόν είναι κάτι πολύ σημαντικό για τη συμπερίληψη των νέων, προκειμένου και οι νέοι να γίνουν ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασία. Αποτελεί τμήμα μια ποιοτική εκπαίδευση και ενισχύει την αποσχολησιμότητα. Η άτυπη και μη τυπική εκπαίδευση είναι επίση πολύ σημαντικά στοιχεία ε, τη διαβίου μάθηση. είναι απαραίτητα εργαλεία για την ε, αντιμετώπιση προκλήσεων όπως είναι η ανεργία. Το Erasmus Plus είναι ένα επιτυχές ε, πρόγραμμα, όμως όλες οι ευκαιρίες δεν έχουν ακόμα αξιοποιηθεί στο έπακρον. Έτσι, θα πρέπει να δοθούν περαιτέρω κίνητρα για τέτοιου είδους ε, κινητικότητα στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, γιατί αυτό θα αυξήσει την απασχολησιμότητα, όπως ε, προκύπτει και από μελέτες της αγοράς εργασίας. Χρειάζεται μεγαλύτερη συνέργεια, λοιπόν, μεταξύ της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας. Κυρία Ντάλτσιλα, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η εκπαίδευση είναι το θεμελιώδες εργαλείο όλων των πολιτών ανεξάρτητα από που προέρχονται. Όλοι θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν στα προγράμματα και στις πρωτοβουλίες για να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Το Erasmus Plus μας βοηθάει ως προς την κινητικότητα και τα κράτη-μέλη μαζί με την Κομισιόν θα πρέπει να εγγυηθούν την ίση πρόσβαση στην κινητικότητα για όλες ε, τις κατηγορίες ανθρώπων, ανεξάρτητα από το φύλλο, για να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση σε όλα τα εκπαιδευτικά και τεχνικά προγράμματα θα πρέπει να μειωθεί το γλωσσικό φράγμα και να λειτουργήσουν καλύτερα τα προγράμματα κινητικότητας για τους νέους και το διδακτικό προσωπικό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μαριά, παρακαλώ ένα λεπτό. Yes, you, Mr. Κύριε Μαριά. Just you. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε ήδη από τον ιανουάριο του 2014 το πρόγραμμα erasmus αποτελεί το νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης το οποίο με προϋπολογισμό δεκαπέντε δισεκατομμύρια ευρώ θα προσφέρει μέχρι το 2020 σε τέσσερα εκατομμύρια φοιτητές τη δυνατότητα σπουδών ή εργασίας σε άλλο κράτος μέλος της ένωσης. παράλληλα στόχος του προγράμματος είναι να βελτιώσει τις προοπτικές σταδιοδρομίας και να παρέχει στους φοιτητές κοινωνικές διασυνδέσεις ωστόσο η κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα καταδεικνύει την ανάγκη αυτό το πρόγραμμα να προσαρμοστεί στι οικονομικέ ανάγκε κάθε χώρα. συγκεκριμένα στι χώρε τη Ένωση παρατηρούνται ακραίε ανισορροπίε στα ποσοστά ανεργία με την ελλάδα να εμφανίζει ποσοστό ανεργίας 24% και ποσοστό ανεργία των νέων 48,9% σαν αποτέλεσμα τη βίαιης δημοσιονομική προσαρμογή και των πολιτικών λιτότητα και μνημονίων που επιβλήθηκαν στην ελλάδα είναι επομένως αναγκαίο η ευρωπαϊκή ένωση να διαθέσει περισσότερα κονδύλια στις χώρες που πλήττονται από υψηλά ποσοστά ανεργίας. ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, Αγαπητοί συνάδελφοι, στην Επιτροπή Πολιτισμού και Εκπαίδευσης εγκρίναμε την έκθεση Μαρακάλ. Γι' αυτό μας κάνει εντύπωση γιατί προβάλλει μια τροπολογία για ένα θέμα που είχαμε απορρίψει στην Επιτροπή. Πιστεύω ότι το θέμα που θίγει, δηλαδή η μετάφραση των εγγράφων, δεν είναι ένα ε, ουσιαστικό πρόγραμμα. Θα πρέπει να υπάρχουν τα κατάλληλα ε, κονδύλια, γιατί θεωρώ ότι είναι μεγάλο γραφειοκρατικό άχθος αν ε, μεταφράσουμε αυτά τα έγγραφα σε όλες τις γλώσσες. Γιατί νόημα έχει να μαθαίνουν και ξένες γλώσσες, όχι να παραμένουμε στις επίσημες γλώσσες σε όλες τους τις εκφάνσεις. Ε, Ιζαμπέλα Ντενόλφη, επίσης για ένα λεπτό. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Η έκθεση έχει θετικές ε, πτυχές, αλλά υπάρχει διστακτικότητα αντιμετώπισης της ανεργίας των νέων. Ιδιαίτερα στη Νότιο Ευρώπη οι δείκτες είναι αποθαρρυντικοί. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη αυτό το χάσμα που υπάρχει, ιδιαίτερα για τους νέους. Πολλοί από αυτούς εγκαταλείπουν και το σχολείο. Γι' αυτό θα πρέπει να μιλήσουμε για αυτό το κοινό αγαθό που θα πρέπει να, στο οποίο θα πρέπει να έχουν πρόσβαση οι πάντες και τα αμαία. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει ίση πρόσβαση και στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης. Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε στη λιτότητα, ιδιαίτερα για τη Νότια Ευρώπη. Ορισμένα μέσα όπως το Ταμείο Εγγύησης των Νέων δεν τα κατάφερε. Η Ευρώπη θα πρέπει να κάνει περισσότερα για, την, για τους νέους. Κυρία Τινόλφη, ο κύριος ο εισηγητής έχει μπλε κάρτα, τη δέχεστε. Όχι, όχι, δεν είναι μπλε κάρτα. Απλώς θα ήθελα να της απαντήσω. Να απαντήσω στην κυρία Χιμένες. Ναι, αλλά είναι πολύ αργά, λυπάμαι. Και προχωράμε στο Καρσιάι. Ντομινίκ Μπίλτ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η έκθεση για το Erasmus Plus είναι μάλλον ικανοποιητική και χαίρομαι που ο συνάδελφος σε ρεαλιστικές προτάσεις που είχα και εγώ προσπαθήσει να υποβάλω σε επίπεδο επιτροπής και κυρίως την ανάγκη να στηριζόμαστε στα επιμελητήρια και τα τεχνικά, τα, τα σώματα των επαγγελματιών προκειμένου να διευκολύνουμε αυτή την κινητικότητα. Βέβαια πρέπει να επισημάνω ότι η διενίσχυση κινητικότητα δεν μπορεί να περιορίσει από μόνη τη την ενεργεία των νέων κυρίω και πρέπει να ληφθούν προκαταβολικά άλλα μέτρα τη κοινή λογική. Πρέπει παραδείγματι να προσαρμοστούν στι ανάγκε τη αγορά εργασία ή θύματα. οι θυματα Η απόκτηση θεμελιωδών γνώσεων, παραδείγματι, η τελευταία έκθεση του Συμβουλίου και της Επιτροπής σε σχέση με το στρατηγικό πλαίσιο 2020 δείχνει ότι μεγάλο ποσοστό των νέων κάτω των 15 έχουν, ελάχιστα, έχουν τεράστια προβλήματα στα μαθηματικά και ένα 18% έχει προβλήματα ακόμη και αναλφαβητισμού στην Ευρώπη. Βεβαίως πρέπει να έχουμε μια διακυβερνητική συνεργασία ευφυή και αποτελεσματική. Η εκπαίδευση όμω είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Παρά τα κενά, η Πρόεδρος, έχετε εξαντλήσει το χρόνο σας και σας ευχαριστώ. Κυρία Σόιντροβα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι πως το Erasmus, το Erasmus Plus είναι ένα από τα κύρια εργαλεία για την επιτεύξη των κοινών μας στόχων, ο περιορισμό της ανεργίας, της φτώχειας, η βελτίωση των ευκαιριών για τον καθέναν, για το κάθε νέο που μπορεί έτσι να έχει υψηλή ποιότητα εκπαίδευση. Η έκθεση αυτή νομίζω στις επαρχές αυτής της βουλευτικής περίοδου είναι επικοδομητική και επικριτική ταυτόχρονα Πρέπει να προσαρμοστούν λοιπόν καλύτερα τα προγράμματα και οι προτεραιότητα. Κύριε Επίτροπε, θεωρώ ότι κλειδί για μια υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης είναι ο δάσκαλος και τα κίνητρα του μαθητή. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προσαρμόσουμε τα προγράμματά μας στην ε, πρακτική εφαρμογή, στην επιχειρηματικότητα, στις ε, γλωσσικές γνώσεις και βέβαια πρέπει να τη διευκολύνουμε και διοικητικά. Ευχαριστώ, όλοι, η Πρόεδρος. Τώρα βλέπω ένα κάποιο, μια κάποια σύγχυση στον κατάλογό μου. Θα ακούσουμε ακόμη, όχι μόνο από τους αριστερές δημοκρατικούς, αλλά και από το ECR και την ALDE ομιλητή. Από τις άλλες ομάδες δεν είχε στήσει κανείς το λόγο. Ε, και έτσι δίνω το λόγο στην κυρία Τσουλιβού για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Με μεγάλη χαρά βλέπω αυτή την έκθεση γιατί πριν μπω στην πολιτική, εγώ ακριβώς αυτό έκανα. Δούλευα με τους ε, νέους ακριβώς για να ενισχύσω αυτού του είδους ε, την ανταλλαγή εμπειριών και σκέψεων με νέους που δεν είχαν τη δυνατότητα και την ευκαιρία να μπουν σε αυτά τα προγράμματα όπως είναι το Erasmus Plus ε, που είναι της τριτοβάθμιας εκπαίδευση. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό που θέλω να σας πω. Το καλοκαίρι του 2014 Ήθελε να συμπαρασταθώ σε ορισμένου ε, και συνεργάστηκα μαζί του. Ε, νέοι λοιπόν, από το Ηνωμένο Βασίλειο, Ρωσία, Ουκρανία και άλλε χώρε. Και για δύο εβδομάδε εργάστηκαν από κοινού στο πλαίσιο του προγράμματο Εράσμου. Και μάλιστα στην περίοδο που υπήρχε πόλεμο μεταξύ Ρωσία και Ουκρανία. Και έτσι αυτοί οι νέοι είδαν πώ είναι ε, και οι άλλοι νέοι από τι άλλε χώρε, παρότι υπάρχει πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών και αυτό δείχνει πώ μπορούμε να ε, βελτιώσουμε την συμβίωση μεταξύ των λαών. Ευχαριστώ κύριε Τοματσίτση για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Το Erasmus Plus είναι ένα σημαντικό πρόγραμμα γιατί προσφέρει ευκαιρίες ε, στους πολίτες που θέλουν ε, να ανοίξουν νέες διόδους, να ερευνήσουν νέα περιβάλλοντα, να αποκτήσουν γνώσεις για τις επιχειρηματικές πρακτικές, μαθαίνουν ξένες γλώσσες, γίνονται έτσι πιο ανταγωνιστικοί στην διεθνή αγορά εργασίας και δεν ε, περιορίζονται έτσι μόνο στην τοπική αγορά εργασίας. Αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να γίνει πιο προσβάσιμο. Να ενισχύσουμε την συμβατότητα μεταξύ των επιμέρους ε, συστημάτων ε, επιστοποίησης και κατάρτισης. Θα πρέπει να δώσουμε πρόσβαση σε αυτά τα προγράμματα σε όλους ε, τους πολίτες, αλλά να μην επιβαρύνουμε αυτά τα προγράμματα με ιδεολογικά στοιχεία και να μην κάνουμε διακρίσεις κατά των ε, μειονοτήτων, γιατί έτσι χάνεται το νόημα. Ευχαριστώ ο κύριος Ναυρατσής και πάλι. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη. Διακόπτη Πρόεδρο, συγγνώμη. Ξέχασα τον τελευταίο μιλητή. Ζητώ συγγνώμη. Γιάνκοφτσιτς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να επισημάνω ότι το Erasmus Plus είναι ένα από τα εξαιρετικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ακούσαμε ότι υπάρχουν και κάποιες ε, δυσκολίες ε, στην υλοποίηση του προγράμματος σε κάποιες περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά έχει βοηθήσει τους νέους να αποκτήσουν νέες δεξιότητες. Θα ήθελα όμως να τονίσω ότι απαιτείται μεγαλύτερη συμβατότητα των ε, προγραμμάτων κατάρτιση των εκπαιδευτών και καθηγητών και αυτό, αυτή η διάσταση θα πρέπει να ενσωματωθεί στο πρόγραμμα. Σε αντίθεση με τον προλαλήσαντα, θεωρώ ότι το τμήμα του προγράμματος ε, που αφορά τις ε, μειονότητες στην Ευρώπη είναι ένα πολύ σημαντικό τμήμα για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ε, ταυτότητας, η οποία υπάρχει είτε μας αρέσει είτε όχι. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα όντως να δώσουμε το λόγο στον Επίτροπο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την έκθεση για το Erasmus για άλλα εργαλεία για την ενίσχυση τη κινητικότητα σε ένα πλαίσιο τη διαβίου μάθηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μαραγκά, τον εισηγητή, για την πολύ καλή δουλειά που έκανε. με την άποψη που αναφέρεται στην έκθεση ότι οι υποτροφίες ε, κατάρτισης και εκπαίδευσης που χορηγούνται από το πρόγραμμα Erasmus ε, αυξάνουν, μάλλον οδηγούν σε απόκτηση νέων δεξιοτήτων, αυξάνουν την απασχολησιμότητα και όλα αυτά τα στοιχεία που αναφέρθηκαν. Για πολλούς τέτοιους μαθητευόμενους, Βλέπουμε ότι η εμπειρία τους από το πρόγραμμα Erasmus Plus είναι η πρώτη ευκαιρία που έχουν να φύγουν από την πατρίδα τους και να μπουν σε μια νέα πραγματικότητα. Η έκθεση Μαραγκάλ συμπεριλαμβάνει μία πλουσιότατη ανάλυση και των ε, πλεονεκτημάτων αλλά και των προκλήσεων της κινητικότητας. Πολλά είναι τα υπέρ. Όταν οι μαθητευόμενοι και καταρτιζόμενοι πηγαίνουν στο εξωτερικό, αποκτούν νέε επαγγελματικέ δεξιότητε που συμβάλλουν και στην κατάρτιση στην πατρίδα του. Επιπλέον, αυξάνεται έτσι και η αυτοπεποίθησή του, ε, προσαρμοστικότητά τους, καθώς και οι δεξιότητες σε ό,τι αφορά οι γλωσσικές, διαπολιτισμικές και το καθεξής. Όλες αυτές οι δεξιότητες που αποκτούν στο εξωτερικό τους δίνουν πλεονεκτήματα για την εσωτερική αγορά εργασία. Οι προκλήσει είναι η έλλειψη χρηματοδότηση ε, γλωσσική και πολιτισμική φραγμή, η χαμηλή συμβατότητα με προγράμματα κατάρτισης στην πατρίδα του μαθητευόμενου, ε, αλλά και διάφορα άλλα νομικά προσκόμματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίγνωση αυτών των προκλήσεων. Θα προσπαθήσω να απαντήσω ε, σε ορισμένα από αυτά τα ζητήματα στον λίγο χρόνο που μου διατίθεται. Η Κομισιόν έχει ήδη διαμορφώσει ένα οργανωτικό πλαίσιο, ε, ούτω ώστε να αυξήσει τι δυνατότητε επιτυχίε του προγράμματο. Η χάρτα κινητικότητα Erasmus Plus, για παράδειγμα, αυξάνει την ε, ενίσχυση ε, των φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και βλέπει και διάφορες στρατηγικές διεθνούς αξιοποίησης αυτών των προγραμμάτων. Να αυξήσουμε λοιπόν την διασύνδεση και με την ε, τοπική αγορά εργασία, ε, να εντοπίζουμε τις κατάλληλε επιχειρήσεις και το καθεξής. Έχουμε και ένα ικανό αριθμό ε, διαμεσολαβητών εντό όπω είναι τα εμπορικά επιμελητήρια, διάφορε ενώσει και τοπικέ αρχέ που βοηθούν στην αύξηση τη ποιότητα αυτών των προγραμμάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα θεωρεί ότι και ιεραρχεί ως προτεραιότητα την αύξηση ε, της δυνατότητας ε, πρόσβασης σε αυτά τα προγράμματα. Καλύπτουμε ακόμα και δαπάνες κατά τη διάρκεια της ε, διαμονής του εξωτερικού. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την απλουστευμένη πρόσβαση στο πρόγραμμα, τα πληροφοριακά μέσα του Erasmus Plus επικαιροποιούνται συνεχώς ε, και κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να απλοποιηθεί η διαδικασία. Σε ό,τι αφορά τις εθνικές αρχές που επεξεργάζονται και αυτές τις αιτήσει, προσπαθούμε να τις ε, συνδράμουμε για να απλουστευτεί η διαδικασία κατά το δυνατόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται ε, στενά και με τις εθνικές αρχές για να υπάρχει ως δυνατόν μεγαλύτερη προβολή αυτών των επιμέρους δράσεων και με εκστρατείες ε, ενημέρωσης σε εθνικό επίπεδο που έχει ως στόχο, για παράδειγμα μία που κάναμε, μια καμπάνια ήταν, ε, είχε ως στόχο να αυξήσει τον αριθμό των επιχειρήσεων που συμμετέχουν. Τέλος, γλωσσική προετοιμασία. Το να γνωρίζει κανείς τη γλώσσα της χώρα υποδοχής είναι πραγματικά κρίσιμη σημασία στοιχείο, ιδίως για νέου μαθητευόμενους που συνήθως ε, δεν έχουν τη γνώση αυτής της ξένης γλώσσας. Εμείς προσφέρουμε επιγραμμικά μαθήματα ξένων γλωσσών και διάφορα άλλα μέσα προετοιμασία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίση συμβάλλει στην βελτίωση τη ε, ε, ποσότητα και ποιότητα τη ε, κινητικότητα. Επομένω, τα προγράμματα και του κύριου Μαραγκαλ και του κύριου Αλτιου, θα δώσουν πολύ σημαντικά χρηματοδοτικά μέσα για την βελτίωση των προγραμμάτων στο μέλλον. Αυτά συνάδουν και με τις προτεραιότητές μας για την ενίσχυση της επιγραμμική εκμάθησης και τη παροχή καλύτερων ευκαιριών στου νέου στην αγορά εργασία. Κλείνοντα, θα ήθελα να πω ότι χαιρετίζω ιδιαίτερω ε, τη δέσμευση του, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αυξήσει την ποσότητα και ποιότητα των προγραμμάτων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Και η Κομισιόν ε, προ την ίδια κατεύθυνση εργάζεται και προσβλέπω σε αγαθή συνεργασία για αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ. πολύ.